Συνάδελφοι, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής πρόοδο στη μεταγωγή κρατουμένων στο Γουαντανάμο και κλείσιμο του Γουαντανάμο. Πρώτα θα ακούσουμε το Συμβούλιο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως τα γνωρίζετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκάλεσε ικανοποίηση η υπόσχεση του κυρίου Ομπάμα, του πρόεδρου Ομπάμα να κλείσει το Γουαντάναμο και αυτό το έκανε όταν έλαβε τα καθήκοντά του. Και υλοποίησε την υπόσχεσή του με εκείνη την κοινή δήλωση. Κοινή δήλωση είπα Ευρωπαϊκή Ένωση 15 Ιουνίου πέρσι. Και με τη σειρά μας. Είμαστε υπέρ του να ισχύσει ο νόμος, το δίκαιο και να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε και είπα σε αυτή την ε, δήλωση θεώρησαν ότι υπ' αυτού του όρου του δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι δεδομένο να υπάρχει αυτό το κέντρο κράτησης και φυλάκιση. Οπότε και στη συνέχεια αυτό ήταν κάτι σαν επιχείρημα, επιχείρημα προπαγάνδας και πρόφαση που χρησιμοποίησε και επικαλέστηκε και επικαλεί το πριν η Αλκάιντα. Πέρασαν χρόνος γιατί υπάρχουν κάποιες δυσχέρειες. Οπότε και ενδεικτικά σας αναφέρω σαν δυσχέρειες ε, σε σχέση με κάποιους κρατούμενους στην Ιεμένη που δεν ήταν δυνατόν να επαναπατριστούν αμέσως, αλλά βεβαίως είναι πολύ καθόδε αυτό το ζήτημα. Είναι επίμαχο, είναι διφορούμε ακόμα και μέσα στη ΣΥΠΑ. Πάντω, εμεί δεν μπορούμε να κερδίσουμε το γεγονό ότι η κυβέρνηση και ο ίδιο ο πρόεδρο συνεχίζουν αυτή τη γραμμή πλεύση για να κλείσουν το Γουαντάναμο. Παρά τη λυσόδια αντίδραση που συναντούν Ακόμα και μέσα στο Κογκρέσο. Ακόμα και μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα και μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Πάντω. έχουμε κάποιους εκεί κρατουμένου οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί στα τακτικά αμερικανικά δικαστήρια. Τζαλίντ Σέιχ Μοχάμετ είναι ένα παράδειγμα. Είναι κάποιο ο οποίος εκρατείτο ε, κατόπιν της επίθεση 11 Σεπτεμβρίου. Οπότε, εμεί ανέκαθεν στι επαφέ μα με τη ΣΥΠΑ ήμασταν ξεκάθαροι σχετικά με αυτό. Και πρόσφατα είχαμε την επίσκεψη του ειδικού απεσταλμένου των ΙΠΑ στι Βρυξέλλε, του Ντάλφ Ρίντ, ο οποίο ήταν παλιότερα ο αρμόδιο για τι σχέσει ΕΕ ΙΠΑ. Τώρα έχει αναλάβει την υπόθεση του κλεισίματος του μου, οπότε ήρθε στις Βρυξέλλες και έγινε ε, και συνεχίστηκε ε, ο διάλογος αυτές τις τακτικές που με τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη ΣΥΠΑ, οπότε και εμείς διατυπώσαμε το ότι ανησυχούμε ε, και προβληματιζόμαστε όσον αφορά αυτές τις λεγόμενες στρατιωτικές επιτροπές για το ότι συνεχίζεται η ούτω η προσωρινή κράτηση χωρί δικαστική απόφαση και για το ότι έχουμε, δεν, δεν, έχουμε, δεν έχουμε κανένα κατάρρευση τη θανατική ποινή και πρόκειται για κάποιε θέσει κρυστάλλινε και μόνιμε και πάγιε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σχέση με τη ΣΥΠΑ και φαντάζομαι ότι και όσον αφορά τι ε, σχέσει μεταξύ των κοινοβουλίων σε αυτόν τον ε, διατλαντικό διάλογο των νομοθετών και εσεί ε, τι ίδιε αρχέ προωθείτε η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι έκανε ότι έπρεπε σχέση με την συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Διατήρησε τα της κοινή δήλωση που σας προανέφερα. Ήδη υπάρχουν κάποια κρατημήρια τα οποία συμφώνησαν να έρθουν στο εδαφός τους κρατούμενοι του γκαντάναμου. σύμφωνα τα αριθμητικά στοιχεία που έχουμε έχουμε επίσης και την ε, Ελβετία ε, και έτσι τις 16 χώρες οι οποίες έχουν συμφωνήσει. Βεβαίως η απόφαση για το αν θα δειχθεί μια χώρα να κρατούν το Γουαντάναμο είναι χώρα είναι απόφαση που είναι απόφαση της κάθε χώρας μέλους. Οπότε αυτό το οποίο θέλαμε ή λέμε πάντα είναι το ότι θα πρέπει να κλείσουν οι φρές του Γουαντάναμου και επίση πρόκειται για κάτι το οποίο αντιβαίνει στα πιο θεμελιώδη ανθρωπινά δικαιώματα. Και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί, να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση και σε σχέση με τι ε, αποφάσει που σα είπα που είναι οι κυρίαρχε αποφάσει κάθε κρατουμένου σε σχέση με την υποδοχή των κρατουμένων. Έχουμε 242 οι οποίοι ακόμα κρατούνται. 44 εξ αυτών έχουν αποφυλακιστεί. Ήταν 242 όταν έλαβε ο Ομπάμα. Και κλείνω κυρία Πρόεδρε γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τις σχέσεις μας αναφέρθηκε στην κοινή δήλωση και θεωρήθηκε ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Θεωρούμε ότι αυτό προσβεύουν και οι ΙΠΑ. Οπότε και εμείς θεωρήσαμε ότι έγινε στροφή της προηγούμενης παλαιότερης πολιτικής της κυβέρνησης των ΗΠΑ για το Γουαντάναμο. Επίσης, διερευνούμε το πώς θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε κάποιες κοινέ αρχές, η μεν και η Να είναι σημείο αναφοράς για τις προσπάθειες της κοινέ καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και αυτά είναι περιεχόμενα της κοινής δήλωσης. Οπότε έχουμε κάθε συμφέρον να κλείσει η φυλακή του Γαντάναμου. Και χαιρετίζουμε το ότι ο πρόεδρος Ομπάμα υλοποιεί την υπόσχεσή του. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχώς σταθερά ζητούσε το κλείσιμο του Γουαντανάμου, όπως ανέφερε ήδη ο κύριος υπουργό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα πλαίσιο για να υποστηρίσει το κλείσιμο του Γουαντανάμου, πρώτα απ' όλα με την απόφαση 4 Ιουνίου 2009 του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών και του Μηχανισμού Ανταλλαγής Πληροφοριών και κατόπιν με την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κρατών Μελών της και τον ΙΠΑ για το κλείσιμο του Γκαντανάμο της 15ης Ιουνίου 2009. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και η κοινή δήλωση δηλώνουν σαφώς πως η απόφαση για την υποδοχή πρώην κρατουμένων και ο καθορισμός του νομικού καθεστώτος τους είναι υπόθεση και αρμοδιότητα του κράτους μέλους ή χώρας συνδεδεμένη στο Σέγγεν. Και οι κρατούμενοι αυτοί μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μέτρα επανένταξης ε, σύμφωνα με τους ισχυρούς εθνικούς νόμους. Στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης, ο πρόεδρος του Συμβουλίου 16 Ιουνίου πέρσι έγραψε μια επιστολή στο συμπρόεδρο της ε, ειδική ομάδας για το κλείσιμο του Κοντανάμου και σε αυτήν την επιστολή αναφέραμε τις αρχές του Εθνούς Δικαίου που αφορούν το κλείσιμο του Κοντανάμου περιέχονται σαφείς δηλώσεις όσον αφορά δικονομικά δικαιώματα όπως η πρόσβαση δικηγόρου και το τι πρέπει να γίνει με την κράτηση, τη μεταγωγή και την απαγόρευση των βασανιστήριων. Έχουν συζητηθεί λεπτομερώς στο διάλογο για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και το διεθνές δικαίο. Η Κομισιόν θεωρεί πως οι εγγυήσεις αυτές είναι σημαντικές για αυτό τον διάλογο καθώς συνεισφέρουν σε καλύτερη αντίληψη του πώς η καταπολέμηση τρομοκρατίας θα σέβεται το διεθνές δίκαιο και το κράτος δικαίου ειδικά όσον αφορά το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους πρόσφυγες και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όπως αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά της θανατικής ποινής και έχει παρέμβει σε μονομές περιπτώσεις ε, σε τρίτες χώρες και στη ΣΥΠΑ για να αποτρέψει τις εκτελέσεις. Η Κομισιόν θα εξετάσει τα απαραίτητα μέσα σε περίπτωση που επιβληθεί η θανατική ποινία από δικαστήριο των ΗΠΑ ή στρατιωτική επιτροπή. Αναγνωρίζουμε τα βήματα που έχει λάβει μέχρι έχει λάβει μέχρι ο πρόεδρος Ομπάμα και ελπίζουμε να συνεχιστεί η διαδικασία στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Τώρα έχουμε τους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. απ' όλα ο κύριος τι ομιλητέ εκ μερου των πολιτικων ομαδων πρωτα απ ολα ο κυριος σαλαφρανκη για δύο λεπτά εξ ονόματο του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Κύριε Επίτροπε, σα υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί όσον αφορά του φυλακισμένου και αυτό έγινε επανειλημμένα και με την ευκαιρία διαφόρων ψηφισμάτων. Όταν ανέλαβε τα κάθηκοντά του, υποσχέθηκε ότι θα κλείσει το κέντρο κράτησης σε ένα χρόνο από τότε. 22 πρώτου Ήρθε αυτή η ημερομηνία. Όμω ε, πολλέ φορέ ε, είναι πιο εύκολο στην πολιτική να κάνει κανεί υποσχέσει, παρά να στηρεί και όπω ε, ανέφερε και ο κύριο Υπουργό είχαμε τον προσωπικό απεσταλμένο ο οποίο ήρθε, μα επισκέφθηκε, συνάντησε μια σειρά παραγόντων εδώ και εξασφαλίστηκε η συνεργασία ε, όπως το τόνισε ο κύριος Επίτροπος. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση τον είπα. και θα, είπαμε ότι θα συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά σε συγκεκριμένες βάσεις και προϋποθέσεις και συγκεκριμένα ε, θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση ασφάλειας για τα κράτη-μέλη. Σε σχέση με όλα αυτά σας υπενθυμίζω την απόφαση ορισμένων κρατών μελών και της ε, Ισπανίας, της χώρας μου αλλά θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της ε, Προεδρίας. Σκοπεύετε να πάρετε κάποια άλλα μέτρα τόσο ώστε να εναρμονιστεί η, η στάση των κρατών μελών σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν στην Ιεμένη. ή θα είναι η κυρίαρχη υπόψη του κάθε κράτου μέλου, ε, ακριβώ όπω αναφέρθηκε στο Συμβούλιο στερικῶν και Υπουργών Δικαιοσύνη, κάτι άλλο. Οι 100 από 190 περίπου ε, κρατούμε, πήγαν στη χώρα προέλευση ή σε τρίτε χώρε. Σε 40 από του κρατουμένου πρόκειται να απευθύνουν σε τακτικά διαστήρια των ΗΠΑ. Ε, Όμω υπάρχουν άλλοι 50. 50 που δεν θα αποφυλακιστούν. Δεν υπάρχουν επαρκεί αποδείξει για να Παραπάνω στη δικαιοσύνη, όμως από την άλλη μεριά θεωρούνται τόσο επικίνδυνοι που οι Αμερικανοί δεν τους απελευθερώνουν. Ερωτώ Κομισιόν και Συμβούλιο. Τι θα γίνει με αυτούς τους 50 κρατημένους οι οποίοι δεν παραπέμπονται στην τακτική δικαιοσύνη. Η κυρία Γκόμες. Το Γκουαντάναμο είναι δημιουργία της κυβέρνησης Bush. Δεν ήταν δυνατό αυτό όμω χωρίς τη σιωπή και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η Ένωση δρά με τις αξίες της πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια για να κλείσει αυτή η φυλακή. Η Διατλαντική Συμφωνία, η καταπολέμηση τη τρομοκρατία, όλα αυτά συνάδουν έτσι ώστε η αίτηση για την αποδοχή κρατουμένων του Γκουαντάνομο να τύχει κοινή ευρωπαϊκή απάντησης. Καθυστέρησε όμως αυτή και μεγάλες χώρες σύνεργοι του Μπούς που ήταν τμήμα της όλης διαδικασίας της Extraordinary Rendition η Γερμανία, η Πολωνία και οι άλλες μεγάλες χώρες τώρα δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους εναντί της κυβέρνησης Ομπάμα. Αυτό είναι θέμα της κοινή εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη θέση μας με βάση το άρθρο 23 της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Χρειάζεται αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η ότι εκπρόσωπος πρέπει τώρα να προτείνει μια πραγματική ευρωπαϊκή στρατηγική για να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν τον Γκουατάναμο και να εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποστήριξη για την ενσωμάτωση των απελευθερωμένων ατόμων και να σεβαστεί το δικαίωμά τους για την οικογενειακή επανένωση. Η Πορτογαλία, η χώρα μου, πρώτα απ' όλα ε, πρόσφερε τη βοήθειά της στην κυβέρνηση Ομπάμα και ήδη υποδεχόμαστε άτομα τα οποία αδίκως υπέφεραν σε αυτήν την φυλακή του Γκουαντάναμου. Ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους Ιβαρώνη Λάντφορτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμμετείχαν ενεργά σε παράνομες εκδόσεις και κρατήσεις, άλλες στήριξαν, άλλες έκαναν τα στραβά μάτια. Οπότε δεν ήταν κάτι που συνέβη κάπου αλλού, Γι' αυτό και μας ενδιαφέρει το ζήτημα. Βεβαίως οι ευρωβουλευτές εδώ και χρόνια ζητούν το κλείσιμο του Γουαντανάμου, οπότε καλωσορίζουμε την ανακοίνωση του Προέδρου Ομπάμα και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες στο να ξεκαθαρίσει το χάλι που άφησε ο Τζόρτζ Μπούς. Αλλά είναι απογοητευτικό το ότι γύρω στα 200 άτομα κρατούνται εκεί. επίση καλωσορίζουμε τι ομοσπονδιακές δίκε για άτομα όπω ο Χαλίτσεκ Μουχάμεντα. αλλά γιατί δεν έγινε πριν από 8 χρόνια η καλύτερη απάντηση στους τρομοκράτες είναι ποινικέ καταδίκες. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δεχτούν την εγκατάσταση περισσότερων κρατουμένων και για λόγους αλληλεγγύης και για λόγους ενοχής για την συνενοχή τους και βεβαίως θα αντισταθούμε στις κινέζικες απειλές για τους Ουιγούρους. Βεβαίως δεν μπορεί να εγκατασταθούν και στη ΣΥΠΑ και αυτό δεν βοηθάει. Ο δικός μου ψηφοφόρος ο Σάκα Αμίρ, ο οποίος ήταν Βρετανός πολίτης και ζούσε στον Πάτρηση στο Λονδίνο, μετά από 8 χρόνια εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα νομικό κενό στο Γκουαντανάμο και φαίνεται πως έχει γίνει μπαλάκι μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΙΠΑ και ίσως υπάρχει μια συμπεγνία για να πάει στην χώρα καταγωγής του, τη Σαουδική Αραβία και είναι άμεσος μάρτυρας των βασανιστήριων που υπέστη ο ίδιος και άλλοι από Βρετανούς και Αμερικανούς πράκτορες. Οπότε μάλλον γι' αυτό δεν έρχεται να καταθέσει τα Βρετανικά δικαστήρια. Καλωσορίζουμε όπως είπαμε τις προσπάθειες να κλείσει τον Κουαντανάμο αλλά είμαστε κατά των στρατιωτικών δικαστηρίων και των λοιπόν παραβιάσεων. Αλλά πρέπει και η Ευρώπη να κάνει περισσότερα. Για τους πράσινους, με συγχωρείτε, η κυρία Χάουταλα για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, αναφερθήκατε στον, στον, εκπροσώπων των ΙΠΑ, οι οποίοι συναντιόνται και με ευρωβουλευτές. Βεβαίως, τα το Συμβούλιο μπορεί να ενθαρρύνει μια κοινή προσέγγιση των κρατών μελών για το κλείσιμο του Γκουαντάναμο. Είναι ξεκάθαρο ότι το Γκουαντάνομο εξακολουθεί να είναι ένα σύμβολο αδικίας και είναι συμφέρον μας να κλείσει. Σήμερα το απόγευμα εκφράζουμε μία άποψη την οποία τακτικά εκφράζει το Κοινοβούλιο μέσω ψηφισμάτων και αποφάσεων. Έχουμε πει στους Αμερικανούς ότι δεν θέλουμε απλώς να μιλήσουμε για την μεταγωγή των κρατουμένων του Γκουαντανομό, αλλά θέλουμε να συζητήσουμε με τις ΗΠΑ και για την πολιτική τους σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις και το κράτος δικαίου. Ελπίζω ότι η φυστάμενη Προεδρία θα, του Συμβουλίου θα έχει τέτοιου είδους συζητήσεις με τη ΣΥΠΑ μέσω του Διατλαντικού Διαλόγου. Τέλος Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η Ευρώπη πρέπει επίσης να ρυθμίσει και τα του οίκου της για τις παράνομες κρατήσεις. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δείξει φως για στον ρόλο των κρατών μελών σε αυτή την παράνομη κράταση. Ο κύριος Γιάννα Τσαρνάσκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπό το φως ε, αυτών των οποίων μόλις είπε η κυρία Χάουταλα αισθάνομαι την ανάγκη να πω πως δεν υπάρχουν στοιχεία στιβαρά που να αποδεικνύουν την ύπαρξη μυστικών εγκαταστάσεων κράτησης τουλάχιστον στην Πολωνία. Όσον αφορά τώρα το θέμα του Κοντανάμου. Είναι σημαντικό το ότι μιλάμε βεβαίως για αυτό το ζήτημα επί κυβερνήσεως Ομπάμα. Νομίζω πως μπορούμε σαφώς να δούμε πως ε, δεν είναι μόνο τμήμα της φρικτής πολιτικής του George Bush ε, του νεότερου. Είναι ευρύτερο το ζήτημα. Το λέω αυτό γιατί ο Ισπανός ε, προεδρεύων του Συμβουλίου μίλησε για την τωρινή αμερικανική θέση. Επίσης θα έλεγα κυρίες και κύριοι πως είναι θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για το θε... να μιλήσει για το θέμα των θυμάτων της νομοκρατίας. Θα δεχτείτε μια ερώτηση από την κυρία Χάουταλα. Κύρια Πρόεδρε, αναφέρθηκα απλώς στα λεγόμενα της πράσινης συναδέλφου. Θα αποδεχτείτε μια ερώτηση από αυτήν, κυρία Χάουταλα. Ε, ευχαριστώ. Κύρια Πρόεδρε, ο κύριος ε, Σαρνέσκι ίσως ε, δεν γνωρίζει πως στις 22 Δεκεμβρίου 2009 μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση παραδέχτηκε για πρώτη φορά πως στην επικράτειά της υπήρχε τέτοιο κέντρο κράτησης. Μια επιτροπή του Λιθουανικού Κοινοβουλίου κατέληξε στο ότι λειτουργούσε φυλακή της CIA στη Λιθουανία στο πλαίσιο καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η λιθουανική κυβέρνηση είχε εμπλακεί νομίζω σε αυτή την δήλωση. Θέλετε να ανταπαντήσετε. Σας ευχαριστώ για την ε, παρατήρηση αυτή, αλλά εγώ είμαι Ευρωβουλευτής της Πολωνίας και όχι της Λιθουανίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Σόλτς κατόπιν από την ΚΟΕ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, χαιρετίζω ρητό στο το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Ασχολείται ξανά με το άμεσο κλείσιμο της φυλακής βασανιστήριων του Γκουαντανάμο και συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη να δράσουν αποφασιστικά. Και πραγματικά είναι ζήτημα υπερατλαντικής ε, συνεργασίας. Σχεδόν 200 άτομα από πολλές χώρες ε, κρατήθηκαν εκεί πέρα κατά παραβίαση των συνθήκων της Γενέβης, χωρίς κατηγορία, χωρίς δίκη και υπήρχαν διάφορα βασανιστήρια και ταπεινώσεις. Το ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, μέχρι σήμερα ασκούσαν πίεση και έλεγαν πως θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάνε σε τρίτες χώρες ή στις χώρες καταγωγής τους είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά κρίμα. Θα πρέπει λοιπόν να ξεσκεπάσει η Κομισιόν την συνυπευθυνότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παράνομη κράτηση αυτών των ανθρώπων εκεί πέρα και είσαι τέλος κάποιες σκέψεις. Η χρησιμοποίηση του Γκαντανάμου για τα βασανιστήρια νομίζω παραβιάζει τις αρχικές συνθήκες τις οποίες είχαμε συνάψει με τις ε, ΙΠΑ και θα έπρεπε νομίζω η κυρία Άστον και οι υπόλοιποι να ζητήσουν επιτέλους να μπει τέλος σε αυτές τις πρακτικές. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νατράς για την Ευρώπη της Ελευθερίας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Εγώ προέρχομαι από τα δυτικά Midlands, χώρα από που, τοποθεσία που προέρχεται και ο Ταλιμπάν που κρατείται στο Γκουαντάναμο, Βρετανός υπήρχος. Η κράτηση πάντως ενός ε, αλλοδαπού είναι σε μια άλλη χώρα, είναι ξένη διαδικασία, είναι προσβολή κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαίου. Μπορώ να σας δώσω ένα κατάλογο Βρετανών πολιτών που έχουν έτσι φυλακιστεί και όχι μόνο στα χέρια της ΣΥΑ και αυτής της διαδικασίας έκδοση αλλά σε χέρια κρατών μελών της Ένωσης με βάση το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που δημιουργήθηκε εδώ έγινε στην Ένωση όλα αυτά. Πριν λοιπόν να καταδικάσετε το, της είπα, κοιτάξτε τον καθρέφτη και κοιτάξτε την υποκρισία σας. Για τους ε, μη εγγεγραμμένους, ο κύριος Ομπερμάιερ, για ένα λεπτό ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το κλείσιμο του Κουαντανάμου είναι οπωσδήποτε ένα μήνυμα για το ότι η ΕΠΑ πρέπει να παραδεχτούν ε, και να τελειώσουν την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σλοβακία, Ιταλία και άλλα κράτη-μέλη δείξαν πως είναι διατεθειμένες να δεχτούν ε, πρώην κρατούμενους. Ε, και βεβαίω αυτό χάρη στη Σέγγεν σημαίνει πως θα μπορούσαν να καταλήξουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αλλά πρέπει να ξεχαρίσουμε τρία σημεία. Πρώτον, και αυτό δεν είναι ε, ντροπή κύριε Σούλτς. Πρέπει να δούμε ποιοι από αυτούς τους ανθρώπους είναι ε, κίνδυνο ασφαλεία, να εξετάσουμε τις σχέσεις με το κάθε κράτος μέλος και εκ των προτέρων να ξεκαθαρίσουμε γιατί δεν μπορεί να πάει στην χώρα προέλευσης ο εν λόγω κρατούμενος. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους μεμονωμένους ομιλητές. Πρώτα από το κύριο Σκοέλιο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το Γκουαντάναμο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φάσματα της διοίκησης Μπούς. Παραβίασε διεθνείς συμφωνίες και την σύμβαση κατά των κρατήσεων. Ήταν αυθαίρετο, δεν σεβάστηκε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και άσκησε βασανισμούς. Ο πρόεδρος Ομπάμα σωστά θεώρησε απαραίτητο να κλείσει τον Κουαντάνο για να έχουν ή ξανά την ηθική θέση που έχασαν με τις πράξεις αυτές ο πρόεδρος Ομπάμα έδειξε την αποφασιστικότητά του και την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του κατήργησε τα στρατιωτικά δικαστήρια και ανακοίνωσε το κλείσιμο του Γκουαντάνομα. Δεν είναι εύκολη η προσπάθειά του γιατί δεν συνεργάζεται το Αμερικανικό Κόγκρεσο. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο συζητήσαμε πολύ για τη διατλαντική συνεργασία αλλά πάντα είχαμε θέση κατά αυτής της φυλακής της ντροπή. Το Συμβούλιο διζήτησε με ψήφισμα όλων των Υπουργών Εξωτερικών το κλείσιμο του Γουαντάνεμο. πολλα Πολλά κράτη-μέλη δέχτηκαν να δεχτούν στην επικράτουά τους κρατουμένους από το Γουαντάνεμο. Η απόφαση να δεχτεί κανένα κρατούμενο ή όχι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να ληφθεί με βάση ευρωπαϊκό συντονισμό. Σε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα και ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να είναι πληροφορία που έχουν όλα τα κράτη-μέλη. Θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για την κατάσταση στην Αμερική και σας ρωτώ τι μπορεί να κάνει ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάνουμε. Τι εμποδίζει κατά την άποψή σας την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει αυτή τη βοήθεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μουνής Οι Δύο λεπτά. Ήταν τερατούργημα πλευράς νομικής και ανθρωπιστικής το Γουαντάναμα παράδειγμα προς αποφυγή. Πόσο μονόπλευρα τα τα πράγματα κυβέρνηση Μπού σε σχέση με τη διεθνική κοινότητα, σε σχέση με τι εξωτερικές σχέσεις, περιφρόνηση του διεθνού δικαίου. Επομένω, θα πρέπει να γίνουν πολλά μετά από την τραγωδία τη κυβέρνηση Μπούς και αυτό το κάνει τώρα ο Ομπάμα. Είχε πει πριν από ένα χρόνο ότι θα είναι μια πρώτη αποφάση το κλείσιμο του Γουαντάναμου. Πρόκειται για μια θαραλέα απόφαση. Επομένω, έτσι θα ανακτήσει την νομιμότητα και την αξιοπρέπεια η, κυβέρνηση των ΗΠΑ όσον αφορά τον υπόλοιπο κόσμο τι έγινε στις 22 πρώτου, ε, το υποσχέθηκε, ε, όμως έχουμε ακόμα 22 ε, κρατουμένους ε, και θα πρέπει μέσα να δούμε μέσω αυτής της στρατηγικής ε, σχέσης μας με την έμπρα του Ατλαντικού, να δούμε πώς θα γίνει αυτό, τι θα γίνει, πώς θα αναδεχθούμε τους κρατούμενους, τους φυλακισμένους του Γαντάναμου εμείς, Ισπανία και άλλες χώρες. Γίνεται αυτό σιγά σιγά επί τη βάση εκείνης της ανακοίνωσης που αναφέρθηκε στις 15 Ιουνίου, ούτως ώστε να έχουμε μια, μια συμφωνία πλαίσιο για αυτή την ε, υποδοχή των κρατουμένους. Όμως πρόκειται για κυρίαρχη απόφαση ε, του κάθε κράτους μέλους και άρα θα πρέπει όμως να δούμε πώς ε, θα δείξει την απαραίτητη αλληλεγγύη Ευρωπαϊκή Ένωση όλοι μαζί. Κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές και, και κυρίως οι σοσιαλδημοκράτες. Είναι 50 οι κρατούμενοι οι οποίοι θεωρείται ότι μπορεί να αποφυλακιστούν ε, και ε, θα πρέπει να δούμε πώς 27 θα προχωρήσουν επί τη βάση του Σέγγεν, του Μηχανισμού ανταλλαγή Πληροφοριών να έχουν ε, μία ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών όσον αφορά την καλύτερη πρακτική για την κοινωνική ένταξη των πρώην κρατουμένων. Ένα λεπτό ο κύριος Έχει το λόγο κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους και του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν για την στάση τους όσον αφορά τον Παντανάμο. Το Παντανάμο είναι μια ανομαλία, μια ντροπή ε, από την σύστασή του ήδη και ίσως ε, θα ήταν ε, δυνατόν να δείξουμε κάποια περισσότερη κατανόηση στην αρχή, αλλά ε, όσο συνεχίζεται είναι μια ντροπή για όλους μας, για όλους εμάς που πιστεύουμε σε αξίες όπως ο σεβασμός των ανθρωπινών δικαιωμάτων και η ελευθερία. Σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη, έτυχε εγώ να δω ένα έγγραφο της ε, κοινή ε, δύναμης ε, για τον Κοντανάμο, μιας οργάνωσης δηλαδή, η οποία θα, θα έπρεπε να μας εξοργήσει. Οπότε έχει φτάσει η στιγμή να πούμε στον κύριο μπαμα να κλείσει αυτή η φυλακή και να τελειώσει αυτή η υποκρισία. Ευχαριστώ. Φλότρο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε τα κράτη-μέλη να υποδεχθούν κρατουμένους από τον Κουαντάνομο που είναι αθώοι. Είναι θύματα αυτοί οι άνθρωποι και πρέπει να τους υποδεχθούμε στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Το κλείσιμο πάντως του Γκουαντάνομο δεν τελειώνει το θέμα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΣΥΠΑ ή στην Ευρώπη. Στη ΣΥΠΑ υπάρχει ακόμα η αντικροτική νομοθεσία που επιτρέπει στρατιωτικά δικαστήρια και ε, κράτηση επαπειρό, αλλά στην Ευρώπη υπάρχουν επίσης προβλήματα και δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε στην Ευρώπη. κυρία Οτάλα σωστά μίλησε για την κοινοβουλευτική έρευνα, μίλησε για την Λιθουανία. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν παράδειγμα. Δεν έχουμε ακόμα εξαγάγει τα διδάγματα από αυτές τις παράνομες πράξεις στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Αυτό είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δουλειά του Συμβουλίου. Πρέπει να εξαγάγουμε όλα τα διδάγματα του τι έγινε για τις παράνομες αυτές πρακτικές και οδήγησαν σε συμμαχία με τη ΣΥΠΑ στη δημιουργία του Γκουαντάναμου. Uh, Έχω πολλά αιτήματα με τη διαδικασία Catch the Eye. Θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε και θα το καταφέρουμε αν σεβαστείτε όλοι το ένα λεπτό ομιλία. Κυρία Ντατή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόσφατα μάθαμε ότι το κέντρο κράτησης του Γκουαντάνομο δεν θα κλείσει όπως είχε προβλεφθεί το 2010 αλλά ούτε καν πριν το τέλος της θητείας του Πρόεδρου Ομπάμα. Το κλείσιμο καθυστέρησε αλλά τουλάχιστον προχωρά. Θα μπορούσε και να είχε διακοπεί. Αυτό είναι και βούληση που έχει εκφράσει η Ευρώπη γιατί δεν μπορούμε χρόνια να κατακρίνουμε τις ΙΠΑ για το κλείσιμο του Γκουαντάναμο και να μην τους βοηθήσουμε για να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα. Πρόσφατα συνάντησα τον Eric Holder, Αμερικανό Υπουργό Δικαιοσύνης, που με εξήγησε το δύσκολο αυτό έργο, αλλά και την βούλησή τους για να έχουν την υποστήριξη των ευρωπαϊκών χωρών για να κλείσουν το κέντρο του Γκουαντάναμο. Υποδεχόμενοι κρατουμένους στην Ευρωπαϊκή Εποκράτεια. Θα πρέπει λοιπόν συντονισμένα να βοηθήσουμε τους Αμερικανούς για να κλείσουν αυτό το οποίο και εμείς ε, θεωρούμε ντροπή εδώ και χρόνια. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Γιατί να υποφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις συνέπειες της αμερικανικής ε, πολιτικής. Ο Αμερικανός ε, πρόεδρος ε, έκανε αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά δεν βλέπω τι σχέση έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άνθρωποι αυτοί απειλήσαν και άλλες χώρες ε, του κόσμου. Βεβαίως είχαμε και τις επιθέσεις, δεν ξέρω αν ξεχάσαμε ήδη το Λονδίνο και τη Μαδρίτη και τα λοιπά τρομοκρατικά χτυπήματα. Είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Θα πρέπει σε αυτή τη φάση λοιπόν πρώτα απ' όλα να δώσουμε το βάρος στην πρόληψη της ε, τρομοκρατίας και να βοηθήσουμε αυτούς τους ε, πρώην κρατούμενους στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία έτσι ώστε να μπορούν να ξαναζήσουν τι τις οικογένειές τους. Ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα, ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισημάνω κάτι που ανέφερε και η κυρία Φλότρ. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε την κυβέρνηση Ομπάμα να κλείσει το Γουαντάναμα γιατί το ζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό και είναι απολύτω απαραίτητο. Θα πρέπει και εμείς ε, να τύχουμε τις δέουσες υποστήριξης και να υποδεχθούμε ε, όσους μας ζητάει η κυβέρνηση Ομπάμα να δεχθούμε αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αν ε, ε, δημιουργήθηκε αυτή η φυλακή είναι επειδή τροφοδοτήθηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό λοιπόν να βοηθήσουμε στο κλείσιμο του Γαντάνομο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη μας για την ύπαρξη, την την ύπαρξη του Γαντάνομο. Γιατί για πολύ καιρό εθελοτυφλούσαμε. Και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όταν ήταν ε, Γάλλος Πρωθυπουργ... Ε, Πορτογάλος Πρωθυπουργός, έδωσε άδεια για υπερπτήσεις των Αμερικανικών ή των αεροπλάνων που περί... μετήγαγαν κρατουμένους και από το Πορτογαλικό έθαφος. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Πρόεδρε, σωστά και όλοι συμφωνούμε να στηρίξουμε έμπρακτα την απόφαση των πολιτειών Αμερικής να κλείσουν το κέντρο κράτησης του γκουαντάναμο και βεβαίω με τα κράτη μέλη της ένωσης να δεχθούν κρατουμένους. Και είναι κοινά αποδεκτό ότι το γκουαντάναμο αποτέλεσε σφάλμα των ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία πρέπει όμω να διασφαλίσουμε ότι τέτοια σφάλματα δεν πρέπει να επαναληφθούν στο μέλλον και δι στην ευρώπη. δυστυχώς όμως έκθεση που θα παρουσιαστεί στο συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του οηε το μάρτιο του 2010, χιλιάδες δέκα προσεχώς δηλαδή εγείρει σοβαρές υποψίες για πρακτικέ μυστικών κρατήσεων υπόπτων και σε κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η μεγάλη βρετανία η ρουμανία και η πολωνία. δεν μπορούμε από τη μια πλευρά να καταδικάζουμε τέτοιε συμπεριφορέ και να λέμε ότι σωστά πρέπει να κλείσει τον γκουαντάναμο και απ' την άλλη να ανεχόμαστε κάποιε αντίστοιχε που ενδεχομένω να πιστεύουμε ότι ίσω να μην συνιστούν τόσο σοβαρό πρόβλημα. όλοι πρέπει να αναλαμβάνουμε τι ευθύνε μα. σα ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αρχίσω από αυτά που είπα Δηλαδή θα πρέπει κατηγορηματικά να πούμε ότι ε, παράνομες φυλακές υπήρξαν και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και στην... Ε, και στη διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Παρόλο που και την Πολωνία δεν υπάρχουν αυτέ οι αποδείξει, υπάρχουν υπόνοιε παρόλα αυτά. Σίγουρα μεταξύ μα δεν υπάρχει καμία διαφωνία ότι θα πρέπει να κλείσει το Γουαντάναμο. Φαίνεται διακυμνού οφθαλμού ότι το θέμα της, ε, του κλεισίματο του Γουαντάναμο θα είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία γιατί δεν υπάρχουν εθελοντέ. Δεν υπάρχουν πρόθυμοι να δεχθούν τους πρώην κρατουμένους. Ερωτώ λοιπόν, έγιναν κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά την, τους μεθόδους κράτησης και ανάκρισης των κρατουμένων, γιατί χρησιμοποιήθηκαν εξευτελιστικές μέθοδοι, απάνθρωπες, κρατούσαν άγρυπνους τους κρατουμένους για, πολύ, για, πολλές, για πολλά μερόνυχτα. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτές οι τεχνικές ανάκρισης έχουν πια καταργηθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Μοβάη. Ευχαριστώ. Και συνάδελφοι, άλλοι όπως και εγώ, είμαστε εξοργισμένοι με τα με τις ε, κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγιναν στο, στο Γουαντάναμο στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση και να ε, δεσμευτούμε ε, να μην υπάρξουν άλλες τέτοιες ε, φυλακές όπως αυτές που υπήρξαν στην ε, Ουγγαρία. Γιατί στην Ουγγαρία έχουμε 12 ε, μέλη της αντιπολίτευσης που βρίσκονται σε ε, κράτηση περιμένοντας δίκη και έχουμε παρόμοιες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν αυτές που έλαβαν χώρα στο Γουαντάναμο. Θα ήθελα οι συνάδελφοι που θέλουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά αυτό το θέμα να σηκώσουν το χέρι και να προωθήσουν μια δράση ε, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα, να ασκηθούν ε, έρευνες. Σηκώστε το χέρι που συμφωνείτε. Καλώς, θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, Προεδρεύοντα να απαντήσει τον εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ. θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πολύ συγκεκριμένα θέματα. Το ένα το επισήμανε ο κύριος Αλαφράκα και το άλλο ο κύριος Σόλτς. Καταρχήν για την Ιεμένη. Από ό,τι ξέρω, για την Ιεμένη δεν υιοθετήθηκε συγκεκριμένη απόφαση για να συνδεθεί η Ιεμένη με κρατουμένους ε, ιεμενικής προέλευσης που βρίσκονται στο Γουαντάναμο. Και μάλιστα το πρώτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα στην ιστορία της Ένωσης για το θέμα αυτό στις 25 Ιανουαρίου, που τακτικό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, κατέληξε σε ένα ψήφισμα όπου ζητούμε πολιτικές ε, και ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις στην Ιεμένη, αλλά δεν γίνεται καμία ανοίξη στο ψήφισμα αυτό για το θέμα του Γουαντάναμο. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση της χώρας αυτής με το Γουαντάναμο. Εμείς υποστηρίζουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, καθώς και τη συνδιάσκεψη που, όπως ξέρετε, έγινε στις 27 Ιανουαρίου στο Λονδίνο. Σε ό,τι αφορά έναν υπενιγμό του κ. Σόλτ για τον κόλπο του Γουαντάναμο και την πιθανότητα να αλλάξει το εδαφικό καθεστώς, αυτό είναι ένα θέμα που απορρέει από μια διεθνή συνθήκη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της ε, Κούβας που ανάγεται στο 1903. Είναι διμερές ζήτημα κουβανικής και αμερικανικής κυβέρνησης. Νομίζω ότι υπάρχει πάντως γενική συμφωνία ότι η φυλακή του Γουαντάναμο αποτελεί ένα χώρο που μαζικά και κατάφορα παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και διατάξεις διεθνούς δικαίου. Και τέτοιο φαινόμενο θα πρέπει να αποτραπεί στο μέλλον. Ασκήσαμε δερμία κριτική εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ύπαρξη του Γουαντάναμο και νομίζω ότι τιμά τον ε, νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών η απόφασή του να κλείσει οριστικά το Γουαντάναμο και μάλιστα να γίνει και μια αναθεώρηση όλης της σοφρονιστικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Η, προ... η... του κυρίου Βάλτς για την εγγενή ανάγκη κλεισίματος αυτής της φυλακής εξαιτίας ε, μαζικής παραβίασης ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι εύλογες όλες αυτές οι παρατηρήσεις και το γεγονός ότι και άλλες χώρες του κόσμου ή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τέτοιε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι δικαιολογία για να αποφύγουμε οποιοδήποτε κριτική. Θα πρέπει να ασκούμε κριτική στην παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου και αναβάνει η χώρα αυτή. Και σα διαβεβαιώ ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμία φυλακή που να μοιάζει έστω και λίγο με τη φυλακή του Γουαντάναμο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εργάστηκαν για το θέμα αυτό και ανέφερα τη διακήρυξη της 15ης Ιουνίου όπου και οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβαν τη δέσμευση να εργαστούν στο θέμα της εμβάθυνσης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαιώματος του αντιτρομοκρατικού αγώνα. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάστηκαν κατάφορα στο Γουαντάναμο. Θα πρέπει λοιπόν όταν γίνεται προσπάθεια καταπολέμηση τρομοκρατία να μην θυσιάζονται στο βωμό τη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με αυτήν την άποψη συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κοέλιο που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να συνεργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρόκειται όμως μόνο για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να κλείσουν το Γουαντάναμα. Γιατί υπάρχουν πολλά συναφή προβλήματα που απορρέουν από το κλείσιμο της φυλακής αυτής και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Άλλωστε ο πρόεδρος Ομπάμα πραγματοποίησε μια σημαντική ρήξη με το παρελθόν. Ουσιαστικά γύρισε τη σελίδα της ιστορίας, όχι μόνο με το Γουαντάναμα, αλλά όλες τις συμπαρομαρτούσε πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο Γουαντάναμα. Και αυτό είναι σαφές και προκύπτει από τις προθέσεις ε, και τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ομπάμα. Για παράδειγμα, σταμάτησαν οι μυστικές κρατήσεις της CIA. Όλοι οι κρατούμενοι συμπεριλαμβάνονται πια στο Διεθνές Μητρό του Έρθρου Σταυρού. Καταργήθηκαν οι βελτιωμένες τεχνικές ανάκρισης της CIA και μάλιστα δεν εφαρμόζονται πια βασανιστήρια ούτε μπορούν να στηριχθούν ε, σε εκθέσεις ε, τέτοιων τεχνικών οι μυστικές υπηρεσίες. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες λοιπόν δείχνουν ότι ο, ο πρόεδρος Ομπάμα πραγματοποίησε μια ρήξη με το παρελθόν και εξέφρασε την προσήλωσή του προς το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Χαιρόμαστε για όλες αυτές τις προϋποθέσεις και το επαναλάβαμε και στην κοινή διακήρυξη. Έγινε μια εις ε, μεταρρύθμιση της θέσης των ε, Ηνωμένων Πολιτειών σε ό,τι αφορά τις ε, πρακτικές ανάκρισης των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, ε, ξανατέθηκαν επιτάπητο στα θέματα της ασφάλειας και αναθεωρήθηκαν με βάση το διάταγμα του, της 27ης Ιανουαρίου του 2009 του Ομπάμα όλα αυτά τα θέματα. Και σίγουρα οφείλουμε να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι φιλοδοξίες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση άσκησε δρυμύτατη κριτική κατά τις φυλακές αυτής και θα πρέπει να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν δύο περιορισμοί. Ένας περιορισμός αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί πρόκειται για θέμα αμερικανικής νομοθεσίας και ισχύει η αμερικανική κυριαρχία για τα θέματα αυτά. Ο δεύτερος περιορισμός είναι ότι και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζουν με κυρίαρχο τρόπο αν θα φιλοξενήσουν, θα υποδεχθούν στο έδαφος τους πρώην κρατουμένους του Γουαντάναμο. Η πρόθεση του Συμβουλίου είναι να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεριμνώντας φυσικά για την τήρηση του δικαιώματος της ασφάλειας στην προσπάθεια του αντιτρομοκρατικού αγώνα. Λοιπόν, συνεργασία, όπως είπε η κυρία Κόμες, είμαστε υπέρ της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπα, αλλά είμαστε υπέρ της συνεργασίας και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των κρατών μέλων. Θα πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας, να έχουμε αμοιβαίο διάλογο και ένα τμήμα του διαλόγου αυτού ξεπερνά το στενό ζήτημα της φυλακής του Γουαντάναμου. Αναφέρθηκε αυτό από πολλούς προλαλήσαντε για παράδειγμα από τον κύριο Σαρνέτσκι, από την κυρία Χαουτέλα. Το θέμα των θυμάτων είναι πολύ σημαντικό και στο διάλογό μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ξεχάσουμε και τα θύματα. Τα θύματα των διαφόρων αυτών εγκλημάτων, τρομοκρατικών εγκλημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει στο μέλλον να το αναλύσουμε. Πάντως σίγουρα θα έχουμε εμβριθεί διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα αυτό. Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι υπάρχει σαφής και κατηγορηματική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα του Γουαντάναμου. Υπάρχει απερίφραστη ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του κλεισίματος του Γουαντάναμου και ξεκάθαρη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά οποιασδήποτε παραβίαση για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για λόγους του τρομοκρατικού αγώνα, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ε, έχουμε την θέληση για αγαστή συνεργασία με τις ΗΠΑ στα θέματα αυτά, γιατί υπάρχει, υπήρξε μια καμπή στην Αμερικανική πολιτική του Πρόεδρου Ομπάμα για το Γουαντάναμο. Και υπήρξε μια ρήξη στο παρελθόν σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική κρατήσεων, τεχνικών ανάκρισης, ε, παράνομα μεταγωγών και ούτω καθεξής. Το Συμβούλιο πάντως θέλει μια συνεργασία με τις ΗΠΑ για να επιτύχουμε το επιθυμητό για όλους που είναι το οριστικό κλείσιμο της φυλακής του Γαντάναμο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος Αμέτσικη. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επαναλάβω ότι κατά τη δική μας άποψη είναι προς όφελος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να κλείσουν οι φυλακές στον Κουαντάναμο. Και όπως είπα και προηγουμένως, η Κομισιόν ε, περιμένει στο μέλλον ε, η Αμερικανική κυβέρνηση να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά αυτό το στόχο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κατά την άποψή μας την ευθύνη για το Κουαντάναμο φέρουν κυρίω σε Ηνωμένε Πολιτείε. Βεβαίω, η Κομισιόν θεωρεί ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί στο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η κυβέρνηση Ομπάμα έχει λάβει κάποια μέτρα, αναφέρθηκαν από τον κύριο Υπουργό απαντώντα στην ερώτηση του κυρίου Ζέμκα, και θέλουμε να πούμε ότι ε, πράγματι ο κύριο Ομπάμα, ο Ομπάμα, ο Ομπάμα, ε, έπαυσε τις ε, τεχνικές ανάκρισεις, κάποιες συγκεκριμένες ε, τεχνικές ανάκρισεις. Ε, απαντώντας τον κύριο Σελαφράγκα, θέλω να πω ότι οι 15 κρατούμενοι, των οποίων δεν έχει αποφασιστεί ακόμα η μοίρα, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε αυτές τις περιπτώσεις και θα καταλήξει σε μία λύση που θα μοιάζει με τις προηγούμενες. Η Κομισιόν δεν έχει λάβει ακόμα την έκθεση της ε, ομάδας κρούσης, ως εκ τούτου και εμείς ε, δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα πιο συγκεκριμένο. Πάντως θεωρούμε ότι ε, θα υπάρξει μια δίκη διαδικασία για όλους. Και τέλος θέλω να σας πω ότι κατά την άποψή μας πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε μια συντονισμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το θέμα αυτό. Και εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόεδρος, έκλεισε λοιπόν τώρα η συζήτηση για το θέμα αυτό ε, και ως εκ τούτου πάμε στο επόμενο θέμα που είναι στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για τις προφορικές ε, ερωτήσεις ε, ε, πρόκειται για την βασική βασικούς στόχου για τη διάσκεψη των συμβαλωμένων μερών της σύμβασης ΣΑΙΤΙΣ. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο